Eh, Καλημέρα σε όλους. Ε, ζητώ συγγνώμη σε όσους ε, περίμεναν εκτός εθούσης, διότι καθυστερήσαμε λιγάκι, σχεδόν μισή ώρα ε, στη συνεδρία των συντονιστών. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω συγγνώμη σε όλους όσους χρειάστηκε να περιμένουν έξω από την αίθουσα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την ημερήσια διάταξη. Καταρχάς Έχουμε την έγκριση της ημερησίας διάταξης. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια αντίρρηση. Εγκρίνεται η ημερησία διάταξη. Στο σημείο 3 έχουμε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίας της 27ης και 28ης Ιανουαρίου 2010. Αν ε, στη διάρκεια της συνεδρίασης δεν υπάρξει κάποια παρατήρηση, θα θεωρούμε ότι εγκρίνονται. Ανακοινώσεις της Προεδρίας. Εξ όσων γνωρίζω δεν έχω τίποτα να σας ανακοινώσω. Να περάσουμε λοιπόν στο σημείο 5. Έκθεση του κυρίου Καντέκ το καθεστώ εισαγωγικών προϊόντων αλληλεία και υδατοκαλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την προοπτική τη μελλοντική μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτική πολιτική. Όπω ε, θα έχετε δει στου φακέλου σα, ο κύριο Κάντεκ παρουσίασε ένα έγγραφο εργασία. Βλέπω ότι ήδη έχει μεταφραστεί σε όλε τι γλώσσε. Ναι, μας επιβεβαιώνει και η γραμματεία, είναι σε όλες τις γλώσσες και το έχετε και στους φακέλους σας. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση λοιπόν, να δώσω το λόγο στον κύριο Κάντεκ για να μας παρουσιάσει το έγγραφο εργασίας. Κύριε Κάντεκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως το είπα ε, και η Πρόεδρος, πρόκειται για ένα έγγραφο ε, εργασίας και όχι για ένα προήμιο ή για μία έκθεση. Είναι ένα θέμα το οποίο ανέλαβα πρόσφατα και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις γιατί αυτό είναι και ο στόχος αυτής της συνάντησης. Ε, αναφερόμαστε σε έρευνες οι οποίες δεν είναι ολοκληρωμένες ακόμη και θα αποτελέσουν τις γενικές γραμμές της έκθεσης. Βέβαια υπάρχουν ακόμη απαντήσεις που πρέπει να δοθούν και περιμένω τα, τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο που έχω απευθύνει. Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να συγκεντρώσω τις ιδέες σας και τις παρατηρήσεις σας και σας καλώ να διατυπώσετε προτάσεις κατά τρόπον ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η έκθεση διότι το έγγραφο αυτό αποτελεί βάση συζητήσεων για σήμερα και θέλω να ακούσω όλες τις αντιδράσεις και ιδίως των σκιωδών ε, ε, εισηγητών αλλά και όλων των συναδέλφων που θα ήθελα να παρέμβουν. Ήδη σε μία πρώτη συνάντηση είχα κάνει μία παρουσίαση ε, αλλά πρόκειται για μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων και έτσι σήμερα προχωρώ περαιτέρω και σας παρουσιάζω τα θέματα που μου φαίνονται ουσιαστικά στην έκθεση αυτή και στο σημείο που βρισκόμαστε τις έρευνες πιστεύω ότι είναι σημαντικά. Είμαι ε, βέβαιος ότι έχετε διαβάσει το έγγραφο εργασίας προσεκτικά. Θα σας υπενθυμίσω όμως τα βασικά θέματα ε, και να θέσω το γενικό πλαίσιο γιατί είναι πολύ βασικό. Ουσιαστικά αναφερόμαστε στην αναδιάρθρωση της κοινοτικής πολιτικής ε, για την ε, αλία και την υδατοκαλλιέργεια ε, στα κοινοτικά ύδατα διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ουσιαστικά μία αγορά που είναι η μεγαλύτερη του κόσμου πριν από τη ΣΥΠΑ ή την Ιαπωνία με πέραν των 300 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2007 και γι' αυτό χρειάζεται αυτή η εκτενής έκθεση διότι σε 8 χρόνια η, η κάλυψη από τους ίδιους πόρους μειώθηκε στο 40% πράγμα το οποίο είναι επίσης ανησυχητικό και αναλόγως των κρατών υπάρχουν διαφοροποιήσεις αλλά αν διαφορε χρησιμοποιήσει κανείς τα αποξηραμένα, τα κατεψυγμένα ε, και νοπά είδη θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ ε, προσεκτικά την κοινοτική πολιτική αλληλείας και υδατοκαλλιέργειας. Ε, δεν, δεν επαρκεί η παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα επαρκέσει και ποτέ στο μέλλον. Υπάρχει απαραίτητη ανάγκη εισαγωγών αλλά παρόλα αυτά πολλοί ε, στο χώρο ανησυχούν είτε για τον όγκο είτε για την τιμή ε, από τις τρίτες χώρες και ιδίως για τις συνθήκες με τις οποίες αλλιεύονται στις τρίτες χώρες και γι' αυτό το έγγραφο αυτό εργασίας εξετάζει όλες αυτές τις πτυχές. Υπάρχουν ορισμένα ουσιαστικά θέματα, δεν θα τα διαβάσω όλα. Υπάρχει μία συνεχώς μειωνόμενη ε, πολιτική της Ένωσης παρόλη την αυξανόμενη κατανάλωση, μία περιφερειακή μειωμένη παροχή η οποία υπάρχει ακόμη, μία κοινή ε, πολιτική η οποία δεν λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των παραγωγών της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι πρόκειται για ένα μη αγροτικό προϊόντα με όλα όσα συνεπάγει και από την άλλη πλευρά ίσως ε, μπορεί να αμφισβητηθεί αλλά από ό,τι έχω ακούσει, από ό,τι έχω διαβάσει, από ό,τι έχω δει, ήδη μπορούμε να σκεφτούμε ότι τα προϊόντα της αλίας και της υδατοκαλλιέργειας σε ορισμένες φορές μπορεί να είναι ένα ε, ε, τρόπος συναλλαγής για, για διάφορες συναλλαγές. Ουσιαστικά η κάλυψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο τελικός στόχος μας και μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην αλληλεία. Υπάρχουν πολλές διαπραγματεύσεις οι οποίες ε, διεξάγονται πολυμερός, διημερός και ε, απαριθμό ορισμένες ε, ή στον ΠΟΕ, η συμφωνία με την Κορέα ήδη, οι ε, διαπραγματεύσεις με τις χώρες Κεντρικής Αμερικής, με τις χώρες των Άνδεων, της ΑΣΕΑΝ, τις ε, διαπραγματεύσεις με τις χώρες Σακέ τις ε, διαπραγματεύσεις ε, με τις Ηνωμένε Πολιτείες και τον Καναδά. Δηλαδή βλέπετε ότι υπάρχουν πολλαπλές διαπραγματεύσεις οι οποίες επίσης είναι ανησυχητικές οι κατηγορίες των εμπλεκομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με συγκρουόμενα κατά ορισμένους χρόνους ε, συμφέροντα ε, οδηγούν ότι άλλοτε τα συμφέροντα ε, συμπορεύονται και άλλοτε, άλλοτε συγκρούονται αναλόγως του είδους που εισάγεται και τις επιπτώσεις στις τιμές δηλαδή αν είναι πολύ φθηνό σε σχέση με το προϊόν τη της κοινοτικής αλληλείας, την ε, ανησυχία για να υπάρξουν ε, οι καλύτερες δυνατές συνθήκες ε, παροχής πρώτων υλών που θα επανεξαχθούν μεταποιημένες, η πορεία του εμπορίου, ο καταναλωτές κακά πληροφορημένοι, οι οποίοι λαμβάνουν αντικρουόμενες πληροφορίες, πληροφορίες και επιπλέον ε, υπάρχουν έχουν ε, και οι επιπτώσεις στις κοινωνικές συνθήκες παραγωγής, ε, στο, στις περιβαλλοντολογικές ε, συνθήκες, οι επιπτώσεις της υδατοκαλλιέργειας και η πληροφόρηση του καταναλωτή. Τέλος, κατά πόσον όλα αυτά αναφέρονται εις την πράσινη βήλο για την αηφόρο ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και αυτό πρέπει να θυγεί στην έκθεση αυτή και από τις πρώτες διαπραγματεύσεις διαπιστώσαμε ότι μπορούμε να, να κάνουμε ορισμένες συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες μπορούν ακόμη να αλλάξουν αλλά υπάρχουν και ε, να αναπτύξουμε ε, την κοινοτική αγορά σφαιρικά και συνολικά για την αλληλεία και την υδατοκαλλιέργεια, να μεταφέρουμε τις αρμοδιότητες για τις διαπραγματεύσεις των προϊόντων αλληλείας και υδατοκαλλιέργειας ε, στον στον ε, Επίτροπο Αλληλείας αντί για τον Επίτροπο Εξωτερικού Εμπορίου που τις διεξάγει τώρα να ε, εξετάσουμε την ε, επίπτωση της αλίες και της υδατοκαλλιέργειας εις τους εμπόρους οι οποίοι ασχολούνται με, αυτή τη, με αυτά τα είδη, ε, να αποφύγουμε κάθε απόκληση από τους κανόνες προελεύσεως για να γνωρίζουμε ποιο είναι το προϊόν το οποίο παραλαμβάνουμε, να υπάρξει μία κοινοτική προτίμηση η οποία να είναι ε, κειμενόμενη αναλόγως των αναγκών, να ε, σεβόμαστε τις ε, υποχρεώσεις μας, να ζητήσουμε να θεωρηθεί ε, το, το προϊόν αλληλείας σαν ένα ευαίσθητο είδος γιατί βλέπετε ότι ήδη που είχε, είχε λεχθεί να ε, σταματήσουν εδώ και τρία χρόνια συνεχίζουν ακόμη ε, να υπάρχει ε, μία σφαιρική αντιμετώπιση των προϊόντων αυτών να απορρίψουμε τις τομεακές αντιμετωπίσεις και να αποφύγουμε τις τεράστιες αγωγές ορισμένων κατηγοριών προϊόντων, να υπάρξει μια κατεπολέμηση του, της παρανόμου αλληλείας ε, να υπάρχει ε, οικολογική σήμανση στα προϊόντα αλίας και υδατοκαλλιέργειας, να ε, υπάρξουν πρότυπα γενικά εφαρμόσιμα και νομίζω ότι πρόκειται για πάρα πολλές προτάσεις τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε. Ένα θέμα το οποίο ακόμη δεν έχω θίξει και μου φαίνεται σημαντικό είναι η, η πτυχή η οποία αυτή τη στιγμή δεν εμφανίζεται στο έγγραφο εργασίας και περιμένω ορισμένε μαρτυρίες από την ακρόαση για να μπορέσω να καλύψω αυτό το σκέλος του εγγράφου. Κατά τα άλλα, πιστεύω ότι από κοινωνικής πλευράς η οργάνωση εργασίας ε, εκφράζει τα κατώτατα αναγκαία πρότυπα εργασίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σέβεται ε, τις ε, συμβάσεις τις οποίες έχει προσυπογράψει και που αυτή τη στιγμή δεν λαμβάνονται υπόψη. Από την άλλη πλευρά, αν εξετάσουμε την ε, κατάσταση του, ε, ε, του ΠΟΕ, πιστεύω ότι χρειάζεται να εξυγχρονιστεί είναι θέμα που έχουμε ξαναθήξει και θα πρέπει και εδώ να αναφερθεί. Και η πρώτη μου κατάληξη, το πρώτο μου συμπέρασμα για συγκεκριμένα θέματα είναι να αναρωτηθούμε αν μπορούμε ακόμη να διατηρήσουμε την ισχύουσα κατάσταση, αν πρέπει να ισχύσει η η ε, ρήτρα της προτιμουμένης χώρας διότι ε, χάνουμε ε, τον τον έλεγχο των προτιμήσεων και δεν θα υπάρχει πλέον η χνηλασιμότης του προϊόντος. Δεν είναι δυνατόν να εξαρτώμαστε από την αλληλεία κατά 70% από την κοινότητα και να αναφέρεται σε ε, τρεις γραμμές ε, εις ε, την πράσινη βίβλο της κοινή γεωργικής πολιτικής και τέλος υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε διότι τουλάχιστον για μένα δεν μπορούμε να θυσιάσουμε ε, το, την Ευρωπαϊκή Αλία στο βωμό των ελευθέρων συναλλαγών. Τεράστιο πρόγραμμα λοιπόν, το οποίο αποτελεί την ε, αρχή των σκέψεών μου, της εργασίας μου, του γράφου εργασίας και τώρα περιμένω από εσά σχόλια για να μπορέσω να το τροφοδοτήσω, να το βελτιώσω. Αντιδράστε, είμαι βέβαιος ότι θα αντιδράστε σε όλα τα θέματα τα οποία έφυξα και τα ε, διάφορα σημεία τα οποία σας επισήμανα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε Καντέκ. Κυρία Ρέιμερς. Καταρχήν, Θέλω να ευχαριστήσω για αυτό το έγγραφο εργασίας το οποίο είναι καλό και αποτελεί ε, ε, μια, μια καλή βάση για το θέμα αυτό. Στο κείμενο λέγεται ότι 60% της ε, έρευνας, της ζητήσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτονται από εισαγωγές. Εδώ λαμβάνονται υπόψη και οι συμφωνίες συνεργασίας και επίσης υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα το οποίο αναγνωρίζω, δηλαδή το εμπόριο με ε, ε, ψάρια για την υδατοκαλλιέργεια που δεν ε, αναλαμβάνεται από την Επίτροπο Αλίας και έχει μικρή σημασία. Ίσως θα έπρεπε να ανατεθεί εις την Επίτροπο Αλίας σε συνεργασία με τον Επίτροπο Γεωργίας. Υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα. Στην παράγραφο που αναφέρεται στην, στο αν συνάδουν οι συμφωνίες να περιλάβουμε και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το οποίο ήδη έχουμε θίξει και τέλος θα ήθελα να πω ότι πρέπει να δεχθούμε τις εισαγωγές γιατί από αυτές εξαρχόμαστε αλλά πρέπει να στηρίξουμε μέτρα κατά τρόπον ώστε να, να στηριχθεί και η δικιά μας παραγωγή και να γίνει και πιο θελκτική. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στίβενσον. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, Αλέν Καντέκ θερμότατα για το πολύ χρήσιμο έγγραφο εργασίας του. Αναφέρατε στην εισαγωγική σας ε, παρουσίαση το θέμα της υγείας και το γεγονός, όπως είπε η κυρία Ράιμερ, ότι για το 60% των αλληλευτικών μας προϊόντων στηριζόμαστε στις εισαγωγές. Και πολύ συχνά ακούμε στην Επιτροπή μας παράπονα ότι δεν υπάρχουν συνθήκες θεμητού ανταγωνισμού. Και το υπογραμμίστε και στην έκθεσή σας, ότι επιτρέπουμε χαμηλότερες προδιαγραφές για τα εισαγόμενα προϊόντα, ενώ είμαστε πιο αυστηροί στις προδιαγραφές που επιβάλλουμε στους κοινοτικούς παραγωγούς. ή στους υδατοκαλλιεργητές. Και πολλές φορές στην Επιτροπή μας ακούσαμε για διάφορα προβλήματα με το Παγκάσιος και το Μεκόν Δέλτα που παρουσιάστηκαν σε μερικές υδατοκαλλιέργειες. Και πολλές φορές ε, οι υδατοκαλλιεργητές ε, μου επισημαίνουν προβλήματα και μου λένε ότι οι Νορβηγοί μετά από πολύ αυστηρές δοκιμές και πειράματα εγκρίνουν συγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα ή συγκεκριμένα προϊόντα για τη χρήση στις υδατοκαλλιέργειες και έχουν έναν απέραντο σχεδόν κλάδο ε, σολομού, καλλιέργεια σολομού. Και εμείς έχουμε αναλύσεις ε, και επιστοποίησεις για τα ίδια προϊόντα στην ε, Ευρώπη. Καλό θα να έχουμε κάποιο συντονισμό με την Νορβηγία, ώστε όταν εμεί εγκρίνουμε ένα προϊόν να μπορούν να το χρησιμοποιούν και οι Νορβηγοί και, το και τα Νάπαλιν. Όταν εγκρίνουν ή πιστοποιούν ένα συγκεκριμένο προϊόν Νορβηγοί, να μπορεί να το χρησιμοποιεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί από τη στιγμή που το χρησιμοποιούν ε, οι Νορβηγοί ευρέω στην υδατοκαλλιέργειά του ένα προϊόν. Οπότε οι αγορέ μα κατακλείζονται από εισαγόμενο σολομό από την Ορβηγία ουσιαστικά δίνουμε στους Νορβηγούς ένα άμεσο ανταγωνιστικό αποτέλεσμα. Ενώ οι δικοί μας επιστήμονες πέραν από πολύ χρονοβόρες και επώδυνες διαδικασίες για να καταλήξουν στην ίδια αξιολόγηση του ίδιου προϊόντος. Ευελπιστώ λοιπόν ότι θα το εξετάσουμε και αυτό το θέμα. Σε ό,τι αφορά την οικολογική σήμανση στην ηχθειοκαλλιέργεια και η δατοκαλλιέργεια και κυρίως να θέσουμε ένα τέρμα στην ανεξέλεγκτη εξάπλωση των ε, ιδιωτικών συστημάτων σήμανσης. Έχουμε, είχαμε ένα τέτοιο παράδειγμα και πραγματικά χρειαζόμαστε μία ετικέτα που θα την εμπιστεύεται το ευρύ κοινό. Οπότε έδωσαν ε, το πράσινο φως σε πάρα πολλά ε, προϊόντα στον κόσμο, το MSC, και ο κόσμος το εμπιστεύεται ως ε, έγκυρο, έγκυρη ετικέτα. Επίσης έχουμε μία σήμανση για τις κονσέρβες τόνου με το Earth Island φιλικό προς τα Δελφίνια σήμα. Και μάλιστα η οργάνωση αυτή λέει ότι αρνείται να βάλει το σήμα της σε κονσέρβες τόνου όταν η εταιρεία αυτή χρησιμοποιεί αυτό το όνομα στο, στην ιστοσελίδα τους και μάλιστα όταν ε, κατά την ε, ε, οργάνωση αυτή, μία οργάνωση δεν τηρεί αυτής αυτέ τι προδιαγραφέ του Dolphin Friend, του φιλικό προ τα δελφίνια, την εκθέτουν στην ιστοσελίδα. Αυτό είναι κάπω αθέμητο ανταγωνισμό. Γιατί μπορεί να είναι φιλικό προ τα δελφίνια ε, μια τέτοια αιλία, αλλά σίγουρα θυσιάζει καρχαρίε, για παράδειγμα ή γονου τόνου. Δεν είναι ότι ε, μια τέτοια σήμανση είναι φιλοπεριβαλλοντική και παρόλα αυτά η οργάνωση αυτή εκβιάζει πολλές ε, ε, εταιρείε κονσερβοποίηση τόνου για να χρησιμοποιήσουν αυτή την σχεδόν απατηλή σήμαση. Γιατί παραπλανεί ουσιαστικά το κοινό ότι επειδή είναι ένα σήμα φιλικό προς τα δεν σημαίνει ότι είναι φιλικό και προ, όλα, προς όλα τα υπόλοιπα αλλιευτικά είδη. Ευχαριστώ κύριε Λέβεν. Ευχαριστώ και ευχαριστώ θερμά και τον κύριο Καντέκ για την καταπληκτική αυτή πρόταση στο άγραφο εργασία του. Γιατί πραγματικά υπογραμμίζει μια σημαντική διάσταση της ελληνικής πολιτικής που δεν αναπτύχθηκε δεόντως στην πράσινη βίβλο και μάλιστα είναι εντυπωσιακό όταν εξετάζουμε τα στοιχεία για το μέγεθος των εισαγωγών και τις διαστάσεις της αγοράς αλίας. Είμαστε η μεγαλύτερη αγορά λευτικών προϊόντων και έχουμε τεράστια επιρροή για τα λευτικά προϊόντα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Οπότε το θέμα αυτό είναι αποφασιστική σημασία. Θα πρέπει να εξετάσουμε τις προδιαγραφέ και τις απαιτήσει που επιβάλλουμε στις εισαγωγέ και να δούμε πώς επηρεάζουν αυτές στο βιωτικό επίπεδο σε ολόκληρο τον πλανήτη. Θα πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί σε θέματα ιχνηλασιμότητας ή την προσπάθεια πάταξης της παράνομης αλίας στον κόσμο. Νομίζω ότι αυτή θα πρέπει να είναι ύψιστη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι όμως που λείπει από το έγγραφο εργασία και συμφωνώ με την κυρία Ρέιμονς, 20% του αλληλευτικού προϋπολογισμού της ε, Ένωσης αφιερώνεται σε αλληλευτικές συμφωνίες με τρίτες χώρες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να δούμε αυτά τα ληφτικά προϊόντα θεωρούν είναι ντόπια παραγωγή ή είναι εισαγόμενα. Είναι αρκετά επίμαχο το θέμα. Επίσης αναφέρθηκε το θέμα των επιχορηγήσεων, των επιδοτήσεων. Να προστατευτούμε από αληφτικά προϊόντα που εισάγονται με συνθήκες dumping στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη επιδοτεί σημαντικά την αλληλευτική της παραγωγή και τον αλληλευτικό της στόλο μέσω αυτών των αλληλευτικών συμφωνιών. Και συνομίλησα με εκπροσώπους ε, αλληλευτικών οργανώσεων της Μαυριτανίας και είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει dumping σε τιμές καλαμαριού για παράδειγμα. Και οι Μαυριτανοί προσπαθούν να ελέγξουν καλύτερα τα πράγματα, να αποτρέψουν ε, την ε, κατάρρευση των τιμών, αλλά ο κοινοτικό αλληλευτικός στόλος συνεχίζει να λιεύει στα μαυριτανικά ύδατα, λες και ήταν ε, χωρικά ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την Ιαπωνία. Θα πρέπει να έχουμε επίγνωση το γεγονός ότι ζητούμε εμείς θεμητό ανταγωνισμό, αλλά δεν τον ακολουθούμε πάντα, γιατί επιβάλλουμε συχνά σε τρίτους κανόνες που εμείς δεν σεβόμαστε. Θα πρέπει και αυτό να το επισημάνουμε στο έγγραφό μας. Ευχαριστώ κύριε Ντότζ. Uh, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και για το έγγραφο εργασίας το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να με υποστεί για λίγο. Το έγγραφο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αν το δούμε πέραν των ε, τρεχουσών συνθήκων ε, κάτω από τις οποίες εργάζονται οι Μίλησα με την ε, βιομηχανία, με τον κλάδο και στην Βόρεια Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο και ένα από τα θέματα που τους απασχολεί ιδιαίτερως στους τελευταίους μήνες είναι η αύξηση των καυσίμων. Πριν από 20 μήνες αυτό κάπως προστατεύθηκε με σχετικά σταθερές ε, τιμές, αλλά η οικονομική πρόγνωση για τους περισσότερους από εμά καταδεικνύει ότι δεν ήταν βιώσιμο κάτι τέτοιο. Επομένως αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ σοβαρή κατάσταση για τους αλληλείς μας. Αν δε το αντιπαραβάλλουμε με το γεγονός ότι το 60% του προϊόντος που χρησιμοποιούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχεται από εισαγωγές, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι αρκετά επικίνδυνη για το μέλλον των αλλιέων. Και νομίζω ότι ο κύριος Καντέκ έχει πάρα πολύ δίκιο όταν μας λέει ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει ακέραιος ο κλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις συνθήκες που ισχύουν αυτή τη στιγμή πόρο απέχει από την πραγματικότητα αυτή. Πολλοί από τις ολίες μας μου λένε ότι οι εισαγωγές έχουν την πιο ε, σημαντική και την πιο μακροπρόθεσμη επίπτωση στην αγορά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική ως προς τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να ε, μπορέσουν να μετριάσουν λίγο τις επιπτώσεις όλων όσων βιώνουν οι αλληλείς. Στόχος όλων μας είναι όχι μόνο να προστατεύσουμε τον κλάδο από τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από τις εισαγωγές, αλλά να ληφθούν και κάποιες αποφάσεις για να αναπτυχθεί ο κλάδος ε, εάν δεν θέλουμε να υπονομεύσουν ε, οι εισαγωγές τη διατήρηση της ε, ζήτησης. Το κείμενο σήμερα το πρωί αναφέρεται και στην υγεία και στα, στις προδιαγραφές παραγωγής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και επισημαίνεται πάρα πολύ ότι χρειαζόμαστε ένα ισότιμο πεδίο για τους αλληλείς μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το είπα και στην Επιτροπή Γεωργίας. Προσφέτως είχαμε το θέμα του βόλου κρέατος από τη Βραζιλία. Ε, είδαμε πώς παράγεται αυτό το βόλιο κρέας και θα ήθελα να επισημάνω στην Επιτροπή μας εδώ σήμερα ότι τα ψάρια δεν διαφέρουν από τη διαδικασία. Θα πρέπει λοιπόν οι μεταποιητές μας να προστατεύονται σε κάποιο βαθμό από εισαγωγές ε, οι οποίες ε, είναι από προϊόντα τα οποία δεν τηρούν τις ίδιες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που τηρούν οι δικοί μας ελίες θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, αυτό για, την, ε, για τον αλληλευτικό μας κλάδο και θα ήθελα πραγματικά να βρίσκεται στο επίκεντρο της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε ο κύριος Φερέιρα. Ε, Ευχαριστώ. Το έγγραφο εργασία του κύριου Καντέκ απαριθμεί μια ευρεία σειρά θεμάτων και από αυτή την άποψη είναι καλό γιατί εντοπίζει σωστά τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και μάλιστα αποτέλεσαν τα προβλήματα αυτά αντικείμενο εκτενέστατη συζήτησης και στην Επιτροπή μας και προτείνει κάποιες λύσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Εκεί όμως θα μπορούσαμε να επικεντρωθούμε καλύτερα στο θέμα της ανέβρεσης λύσεων και σίγουρα το θέμα αυτό θα μπορούσε να το αναπτύξει περαιτέρω ο κ. Καντέπ. Τα προβλήματα τα εντόπισε σωστά, με οξυδέρκεια. Θα πρέπει όμως οι προσανατολισμοί που θα προτείνει να είναι πιο σαφείς και οι λύσεις επίσης ε, πιο απτές. Σε ό,τι αφορά τις ανησυχίε, για παράδειγμα, που δημιουργεί η απελευθέρωση του εμπορίου, όπως ε, εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν διασκεδάζονται όλε αυτέ οι ανησυχίε από την απελευθέρωση του εμπορίου. Θα πρέπει λοιπόν να αντιλήσουμε κάποια συμπεράσματα. Η απελευθέρωση του εμπορίου δεν μπορεί να συνεχιστεί με τον τρόπο που εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα. Και πολλοί συνάδελφοι ανέφεραν την ανάγκη της αξιολόγησης ε, της συγκλασιμότητας ε, των κανόνων προέλευσης Επίσης θα πρέπει να αξιολογηθεί η επίπτωση της κάθε διαπραγμάτευσης, γιατί πολλές φορές οι διαπραγματεύσεις προχωρούν χωρίς να πληρούνται αυτά τα κριτήρια. Έχουν προσδιοριστεί διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, το Μαρό κτλ. που αμελούν τελείως αυτά τα θέματα. Η απελευθέρωση του εμπορίου όπως εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας ικανοποιεί. Και εκεί θα πρέπει να έχουμε μια περίφραστη θέση και κατηγορηματική απόρριψης ε, του τρόπου εφαρμογής αυτής της απελευθέρωσης. Θα πρέπει για να συνεχίσει η απελευθέρωση να υπακούσει κάποιους κανόνες. Μερικοί αναφέρονται, θα πρέπει να τους εμπλουτίσουμε. Επισημάθηκαν επίσης τα αντικρώμενα συμφέροντα ορισμένων φορέων του κλάδου και πολύ σωστά εντοπίζεται αυτή η σύγκρουση των συμφερόντων. Υπάρχει η σύγκρουση αυτή, αλλά καλή διάγνωση. Δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτωχοι σε αυτή τη διαπίστωση. Θα πρέπει να προασπίσουμε τα συμφέροντα των παραγωγών, να διασφαλίσουμε την παραγωγή μας, παρόλο που κάτι τέτοιο σήμερα μπορεί να σημαίνει ότι θα έρθουμε σε αντίθεση, θα διακυβεύσουμε κάποια συμφέροντα των ε, μεγάλων εταιριών διανομής. Θα πρέπει να λάβουμε μια πολιτική θέση απέναντι σε αυτή τη σύγκρουση συμφερόντων και πιστεύω ότι η θέση μας θα πρέπει να είναι υπέρ της προάσπισης ε, των συμφερόντων των παραγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι των διανομέων. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει και κάποιο περιθώριο λιγμών σε ό,τι αφορά την διατράνωση της δυνατότητας και της ανάγκης να αντιστρέψουμε αυτή την τάση αύξησης των εισαγωγών και όλο και μεγαλύτερης εξάρτησής μας από τους εισαγωγείς. Θα πρέπει να αντιστρέψουμε αυτή την τάση, να μειώσουμε κάπως αυτή την εξάρτησή μας από εισαγόμενα προϊόντα. Άλλοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν σε θέματα πιστοποίησης

Θα πρέπει λοιπόν να μεταφραστεί σε συγκεκριμένα χειροπιαστά μέτρα για να αποτρέψουμε αυτή τη θυσία της κοινοτική ελίας στο βωμό του ελευθέρου εμπορίου. Πολύ σωστά, νομίζω και πολύ εύστοχα συνόψε το πρόβλημα ο κύριος Καντέκ. Αυτή η ιδέα πάντως που είναι κέρια θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια και από το έγγραφο και να συνοδεύεται από συγκεκριμένα μέτρα για να εφαρμοστεί. Να αποτραπεί δηλαδή αυτή η θυσία. Ο κύριος Μιλάνα. Ο κύριος Γκόρμπατσεκ ήθελε να μιλήσει και αυτός, ε, συγγνώμη, όμως προηγείται ο κύριος Μιλάνα. Καταρχάς, συγχαρητήρια στον κύριο Καντέκ, διότι κατάφερε να βάλει όλα τα πράγματα στη σειρά τους. Περιλαμβάνονται τα πάντα και πιστεύω ότι ορθώς ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή μας, συγγνώμη, έκανε αυτή την, την γνωμοδότηση ίδιας πρωτοβουλίας, διότι θέτει το πλαίσιο της συζήτησης, της μεταρρύθμισης της κοινής ελευτικής πολιτικής, όπως και η γνωμοδότηση που θα συζητήσουμε σε κάποιες εβδομάδες για τα θέματα της υδατοκαλλιέργειας. Έχω κάποιες παρατηρήσεις, όλες ε, θετικές, καμία ένσταση συγκεκριμένη τουλάχιστον. Καταρχήν, θα πρέπει να κατανοήσουμε τι είναι η ευρωπαϊκή αλία; Ποια είναι. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ εύστοχη η παρέμβαση της κυρίας Λεβίν. Είναι τα ψάρια τα οποία λεύουμε στις θάλασσές μας ή είναι ε, τα ψάρια τα οποία λιώνουν οι επιχειρήσεις μας. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική διευκρίνηση διότι ε, προϋποθέτει και μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Η πρώτη είναι η παραγωγική διαδικασία, η δεύτερη είναι η βιομηχανική διαδικασία με όλες τις, τις ε, επιδράσεις. Ε, πρόκειται για μια δραστηριότητα η οποία έχει πολλές ομοιότητες με την εμπορική δραστηριότητα και για αυτές τις επιχειρήσεις πολλά από τα αλλιεύματα είναι αλλιεύματα τα οποία προκύπτουν από εισαγωγές. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε μία αγορά η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση και κανονικά θα έπρεπε να επιληθεί πλήρως το ζήτημα της ε, τοπικής παραγωγής και εδώ έχετε και η αντίφαση. Πολλές φορές η τοπική παραγωγή έχει ένα ουσιαστικό πρόβλημα και δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική με την ε, ευρύτερη αλληλεία. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη αντίφαση. Σημαίνει ότι υπάρχει μία λανθασμένη ε, πολιτική, η οποία υφέρπει, φαίνεται ότι κάνουμε λάθος και στις εθνικές μας πολιτικές και στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Διότι σε κανέναν άλλο τομέα, όταν υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση, δεν έχει τόσα προβλήματα η τοπική παραγωγή. Και εδώ ακριβώς πρέπει να κάνουμε την παρέμβαση εμείς. Θα πρέπει η ανταγωνιστικότητα αυτή ε, να πάψει να εφίσταται. Και οι ροές παραγωγής θα πρέπει να συσχετιστούν και με τα όρια της παραγωγής. Η, τα στοιχεία κλειδί τα οποία αναφέρθησαν και περιλαμβάνονται στο έγγραφο είναι τρία. Η σήμανση, η χνηλασιμότητα και οι σχέσεις με τον καταναλωτή. Θεωρώ ότι στην έκθεση θα πρέπει να αναπτύξουμε λίγο περισσότερο αυτό το επιχείρημα και αυτό το οποίο περιλαμβάνεται στην έκθεση, δηλαδή το να περάσουμε από το τελευταίο πρόβλημα ε, του εμπορίου και να με το πρώτο πρόβλημα της αλληλείας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η αλληλοσύνδεση με όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Επαναλαμβάνω ότι τρει είναι οι λέξει κλειδί, σήμανση, χνηλοσημάτητα και σχέση με τον καταναλωτή. Θα ήθελα να κάνω και κάποιε προτάσει προ τον κύριο Καντέκ. Επιφυλάσσομαι να του στείλω και κάτι γραπτό, το οποίο θα μπορούσα να του στείλω τι επόμενε μέρε και κάποιες ε, σκέψεις για τα όσα κάνετε. Είμαστε πλέον μία αγορά 12 εκατομμυρίων τόνων αλευμάτων. Τα μισά προέρχονται από την υδατοκαλλιέργεια. Δηλαδή, τα μισό της καταναλώσής μας, 5,5 εκατομμύρια περίπου τόνοι, καταναλώνονται στην Ευρώπη και προέρχονται από την υδατοκαλλιέργεια. Τούτο σημαίνει ότι και το έγγραφο θα πρέπει να έχει αυτό, αυτή τη διτή προσέγγιση. Δηλαδή, υπάρχει μια πολιτική η οποία θα πρέπει να οικοδομηθεί γύρω από το προϊόν που αλλιεύεται από τις θάλασσες και επίσης μια πολιτική που θα πρέπει να οικοδομηθεί γύρω από τα προϊόντα της υδατοκαλοέργειας. Δεν μπορούμε να έχουμε την ίδια προσέγγιση και από πλευράς οικονομικών κύκλων που συνδέονται με τους μηχανισμούς εισαγωγών και εξαγωγών. Διότι και εμείς για κάποια προϊόντα είμαστε εξαγωγές. Παραδείγματο χάρη εξαγωγές ε, σολομού. Ο σολομός δεν παράγεται για να καταναλώνεται μόνο, ε, παράγεται και για την εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, εγώ θα έκανα εδώ τη διάκριση μεταξύ των δύο, διότι δεν μιλάμε ακριβώς για την ίδια πολιτική. Στην πρώτη περίπτωση, θα πρέπει να γίνει μια συντονισμένη εργασία από πλευράς Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο θέμα της ιδετοκαλλιέργειας θα πρέπει να ε, γίνει πολύ πιο συστηματική η παραγωγή και θα πρέπει να δημιουργηθούν πολιτικές ε, για τη σήμαση και την αγνώριση από πλευράς καταναλωτών των προϊόντων. Όσον αφορά τώρα στην παραδοσιακή αλληλεία, δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε την ίδια πρόταση. Δηλαδή, να κάνουμε μια διάκριση για τα ευρωπαϊκά αλλιεύματα, αυτά που αλλιεύονται στην Ευρώπη. Το παράδειγμα που έγινε πριν για τα ζωοτεχνικά μέσα και τα βοηδή από την ε, Βραζιλία, που είναι ένα συγκεκριμένο προϊόν με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω αν υπάρχει γόνιμο έδαφος και για μας ε, για να μπορούμε με κάποιο τρόπο να αναγνωρίζουμε τα προϊόντα μας ως προερχόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα όμως να σταθούμε και σε αυτό. Θα ήθελα να επισημάνω επίσης και τις πολιτικές ε, που αφορούν τους καταναλωτές. Στον τομέα της αλληλείας δεν υπάρχουν πολιτικές καταναλωτή. Ενώ στο εσωτερικό των πολιτικών της κοινή ελευτικής πολιτικής υπάρχουν κανονισμοί, υπάρχουν νοτροπές, υπάρχουν συμπεριφορές οι οποίες μας ε, κατευθύνουν και ρίχνουν το μάτι και προς τον καταναλωτή, φαίνεται ότι εμείς στην Ελία δεν έχουμε δημιουργήσει στρατηγικές που να οδεύουν προς αυτή την άγουσα. Πρόκειται λοιπόν για ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο, διότι στο κάτω-κάτω της γραφής αυτός που επιλέγει είναι ο καταναλωτής. Αυτός που ε, εμπλουτίζει ή τοχαίνει μια περιοχή είναι ο καταναλωτής διότι αυτός είναι αυτός που επιλέγει στην αγορά το τελικό προϊόν. Να ολοκληρώσουμε κάτι που σας είπα ήδη. Θα πρέπει στο επίκεντρο των γενικών κατευθύνσεων της ε, αλίας θα πρέπει να υπάρχει ε, κυρίως ε, το θέμα του, της Αλίας αυτής καθ' αυτής και όχι του εμπορίου. Το επιχείρημά μου, η λογική μου, συνδέει και τα όσα περιεχάμενονται στην έκθεση της κυρίας Πατράους και αυτό που γράφω εγώ στην έκθεσή μου για την υδατοκαλλιέργεια και αυτά που αναφέρονται εδώ στο έγγραφο εργασία. Νομίζω ότι μιλάμε για τρει όψει του ίδιου νομίσματο. Βέβαια, συνήθω ένα νόμισμα έχει δύο όψει. Εμεί όμω έχουμε τρει όψει του ίδιου νομίσματο. Έχουμε και το προφίλ, αν θέλετε. Έχουμε τι δύο όψει και έχουμε και το. Ε, και το προφίλ. Και αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε ιδιαιτέρως. Θα πρέπει να ξεκινήσει μια περίοδος για την Ευρώπη, στην οποία η πολιτική αλληλείας θα είναι ε, ευγενείς όσο είναι και η πολιτική γεωργίας. Θα έχουμε, πρέπει να λάβουμε λοιπόν όλες τις πτυχές υπόψη και θα ήθελα να υπάρχει και αυτή η πιο γενικευμένη έννοια στο έγγραφο εργασία σας. Ευχαριστώ. Θα σας διαβάσω τον κατάλογο των αγορητών. Andrés Barea, η Πατράου η Θέλει άλλος κανείς το λόγο για να κλείσουμε τον κατάλογο. Ο κύριος Πρόβατσεκ. Ευχαριστώ. Γκρέμπερτσικ, συγγνώμη. Νομίζω ότι δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε με αυτά που ακούσαμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα σημεία του εγγράφου εργασία και ευχαριστώ θερμά τον κύριο Καντέκ για το έγγραφο, γιατί πραγματικά είναι κέρια σημασία όλα αυτά τα σημεία που αναπτύσσει. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα θέμα, κύριε Καντέκ. Δυστυχώς αυτά τα, αυτά τα ζητήματα δεν είναι μια απλή διάγνωση, αλλά πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη της μελλοντικής ελευτικής πολιτικής. Είχαμε βέβαια την πράσινη βίβλο και δεν προσθέθηκε τίποτα άλλο, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και το εξής. Αυτό το έγγραφο, αυτό το έγγραφο εργασίας, μπορεί να αποτελέσει δομικό στοιχείο για την οικοδόμηση της μελλοντική αλληλευτικής πολιτικής. Είναι εξίσου θεμελιώδης αυτό το έγγραφο εργασία με την πράσινη βίβλο. Και αν συνδυαστεί με την πράσινη βίβλο θα μπορούσε να μας προστατεύσει από αυτή την αχίλιο πτέρνα που έχουμε στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και που είναι ε, η μαζική εισαγωγή αλληλευτικών προϊόντων. Θα πρέπει να προφυλαχθούμε βέβαια από μια πολιτική dumping που γνωρίζουμε ότι εφαρμόζεται από ορισμένα άλλα κράτη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν στοιχείο και αναπόσπαστο της μελλοντικής ελευθερικής πολιτικής στο έγγραφο. κυρία Αντιβαρέα. Συγχαρητήρια κύριε Καντέκ. Γιατί όπως φάνηκε από τους προλαλήσαντες, το έγγραφό σας είναι ιδιαίτερα αξιόλογο. Και το θέμα που πραγματεύεστε φυσικά είναι νευραλική σημασία και θέσετε το δάκτυλο επί των τύπων των ήλων πραγματικά. Πολλά αυτά τα ζητήματα έχουν χαρακτήρα οριζόντιο και αφορούν όχι μόνο την αλία αλλά και το εξωτερικό εμπόριο, τα αναπτυξιακά ζητήματα, την εξωτερική διάσταση. Είπατε ότι έχουμε πρόβλημα αγοράς. Πολύ σημαντικό. Υπάρχει πρόβλημα αγορά και στη προσπάθεια μεταρρύθμιση αυτή τη κοινή ελληνική πολιτική θα πρέπει να επισημάνουμε το πρόβλημα και να έχουμε υπόψη την ενιαία αγορά και να περιορίσουμε τις επιθέσεις που υφίσταται από εισαγόμενα προϊόντα που οδηγούν σε μια κατάρρευση των τιμών. Βέβαια, βρισκόμαστε σε ένα παγκόσμιο κόσμο, έχουμε εμπορικέ συναλλαγέ, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε εισαγωγέ. Αλλά στι συμφωνίε εισαγωγή ε, που εξετάζουμε θα πρέπει να δούμε τις επιπτώσεις τους ε, το, από εμπορική άποψη, από κοινωνική άποψη, ε, ε, για την απασχόληση, αλλά και από άποψη αναπτυξιακή να γίνει η επιπτώση όλων αυτών των επιπτώσεων, ε, αξιολόγηση συγγνώμη, όλων αυτών των επιπτώσεων μιας συμφωνίας. Επίσης θα πρέπει να αξιολογηθεί η συνέπεια κάθε διαπραγμάτευση και αυτό θα πρέπει να το κάνουμε εμείς στην Επιτροπή μας, γιατί όλες οι συμφωνίες έχουν ένα κοινό κορμό, ένα γενικό, αλλά και ένα, ένα ειδικό τμήμα που συγχαίει τις τρεις πλευρές εμπόριο, εκεί βοήθεια και αλεία. Θα πρέπει όλες αυτές τις πτυχές να τις αναλύουμε στην αξιολόγησή μας για κάθε διαπραγμάτευση και συμφωνία. Γιατί, επαναλαμβάνω, υπάρχουν εγκάρσεις επιπτώσεις και σε καμία περίπτωση θα πρέπει να βρεθεί χαμένη από όλη αυτή την ιστορία η κοινοτική αλεία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Καντέκ για την εξαιρετική του έκθεση και να ζητήσω συγγνώμη που άργησα να φτάσω. Ήρθα από τη Φιλανδία σήμερα το πρωί και ο λόγος για τον οποίο ήρθα σήμερα και όχι εχθές ήταν ότι εχθές ψάρευα, ε, χειμερινή αλληλεία. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο μέτρα πάγο ε, στη θάλασσα, παρόλα αυτά ψαρεύουμε δύσκολα και γι' αυτό εισάγουμε πολύ ψάρι το χειμώνα παίρνετε ένα σιδηροπρίονο, κάνετε μία τρύπα και μπορείτε να ψαρέψετε. Αλλά γι' αυτό εισάγουμε πολλά ψάρια και γι' αυτό η έκθεση αυτή μας ενδιαφέρει πολύ. Ο κύριος Καντέκ έκανε πολύ καλή δουλειά και η έκθεση αυτή αναφέρει πολλά σημαντικά σημεία. Προσωπικά είχα τη χαρά να φάω πολύ ωραίο ψάρι εχθές, διότι αφού ψαρέψαμε φάγαμε τα ψάρια μας και ήταν το καλύτερο ψάρι που φάγαμε εδώ και πολύ καιρό. Είδαμε λοιπόν πόσο καλύτερα ε, ε, καλύτερη γεύση έχει το ψάρι αν το φάτε αμέσως. Ξέρω βέβαια ότι οι καταναλωτές έχουν την ίδια εντύπωση, δηλαδή το ψάρι έχει πολύ ωραιότερη ε, γεύση παρά αν έχει περάσει ώρες στο αεροπλάνο σε μια συσκευασία καινού αέρα και Γι' αυτό πρέπει να προσφέρεται με τον καλύτερο τρόπο το ψάρι αυτό. Ξέρω ότι και η οικολογική σήμανση είναι πολύ σημαντική, ένα θέμα το οποίο πρέπει να τονίσουμε και επίσης νομίζω ότι στο παρελθόν δεν είχαμε ασχοληθεί για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις για την αλληλεία από τρίτες χώρες διότι αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι από πολιτικής απόψεως και πρέπει να ε, εξετάσουμε το θέμα αυτό. Ίσως από πλευρά των βορείων χωρών ε, ορισμένοι μου έχετε πει ότι πάντοτε μιλάμε ε, για τις φώκες και τους κορμοράνους αλλά ε, ο λόγος για τους οποίους θίγουμε είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε ψάρια στη Φιλανδία. Εάν όμως, εάν όμως συντηρούμε και διατηρούμε ε, τις φώκες και τους κορμοράνους που τρώνε πολύ ψάρι πρέπει εμείς ε, να εισάγουμε από την Νορβηγία. Ε, πρέπει να βρεθεί σωστή οικολογική σήμανση διότι οι άνθρωποι θα προτιμούσαν να έχουν ψάρι που ξέρουν από πού προέρχεται και πρέπει να βρούμε μία καλή ισορροπία μεταξύ το, της πολιτικής θελήσεως του Κοινοβουλίου και ε, της... Ε, ε, και των πολιτικών επιταγών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Καντέκ για το έγγραφό του αυτό είναι μια βασική ε, έκθεση κατά πρωτοβουλία για ένα θέμα το οποίο έχουμε εξετάσει ακόμη και ε, αν ε, ε, έχουμε εξετάσει και άλλα πολιτικά προβλήματα και γι' αυτό άργησε πολύ να κοινοποιηθεί αυτή η πρωτοβουλία. Εμένα μου αρέσει η μορφή του εγγράφου αυτού γιατί μπορεί να ε, παρουσιάσει σωστά τα σημεία που απετέλεσαν ε, θέματα συνενέσεως αυτής της Επιτροπής και να τονίζει ότι υπάρχει συνένεση στη συζήτηση ε, και έτσι ο κύριος Καντέκ ε, το αναφέρει και διευκολύνει τη δουλειά μας. Πρέπει να προσθέσουμε μία πρωτοβουλία αλλά τα βασικά θέματα έχουν παρουσιαστεί και αυτό είναι πολύ ουσιώδες. Ε, υπάρχει όμως ένα θέμα το οποίο πρέπει ακόμη να αναφερθεί. Το γεγονός ότι στο τέλος πρέπει να διατυπώσουμε συγκεκριμένες προτάσεις διότι εφόσον υπάρχει συνένεση για όλα αυτά τα θέματα και υπάρχει, τότε θα πρέπει να δούμε ε, πώς θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτά που ζητάμε και να περάσουμε από τις αρχές και τα λόγια στα έργα και στην πρακτική. Σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ ότι τα προϊόντα εχθειοκαλλιέργειας και υδατοκαλλιέργειας και αλίες είναι ευαίσθητα προϊόντα. Συμφωνώ με την διαπίστωση αυτή. Και επειδή συμφωνώ με πολλούς ε, προλαλήσαντες, δεν πρόκειται να επαναλάβω τα σχόλιά τους. Θα ήθελα να επιμείνω σε ορισμένα θέματα που δεν υπογραμμίστηκαν αρκετά. Για παράδειγμα, τα ελληνικά προϊόντα και τα προϊόντα το σε επαναλαμβάνω, είναι ευαίσθητα προϊόντα. Δεν είναι απλώ εμπορεύσιμα αγαθά σα χωρίς ιδιαιτερότητα. Έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αυτή η ιδιαιτερότητα θα πρέπει να αναγνωριστεί για τα λευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργεια. Δεν είναι τυχαίο αγαθό, ένα τυχαίο εμπορικό προϊόν αυτά τα αγαθά. Επίσης είναι τρόφιμα. Θα πρέπει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διατρανώσει τη θέση του ότι αυτά τα προϊόντα δεν είναι απλά εμπορικά αγαθά, αλλά έχουν ιδιαιτερότητα και αυτή η ιδιαιτερότητά τους θα πρέπει να διαφυλαχθεί. Κάτι άλλο που θα ήθελα να τονίσω αφορά την ανάγκη να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη. Προτείνεται η μεταβίβαση της αρμοδιότητας ε, για τις ελληνικές ε, συμφωνίες από το εξωτερικό εμπόριο στην Αλία. Εδώ δεν θα μιλούσα για μεταβίβαση αρμοδιότητων, αλλά περισσότερο για ανάμειξη, γιατί δεν νομίζω ότι μπορούμε να μεταβιβάσουμε αυτές τις αρμοδιότητες ε, από τον αρμόδιο επίτροπο εξωτερικού εμπορίου στην επίτροπο αρμόδια για την Αλία. Γιατί μια τέτοια μεταβίβαση θα μπορούσε κανεί να διεκδικήσει και για πολλά άλλα θέματα. Πάντω πιστεύω ότι ο αρμόδιο επίτροπο για το εξωτερικό, για το διεθνέ εμπόριο, θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την αρμόδια επίτροπο Ελία για τα προϊόντα αυτά. Ανάμιξη λοιπόν, όχι μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. Είναι σημαντικό λοιπόν, μια και μιλούμε για αλλιευτικά και είδα το προϊόντα το καλλιέργεια, να υπάρχει στενή ανάμιξη και συνεργασία Στι συμφωνίε αυτέ μεταξύ του Αρμοδίου Επιτρόπου για το Εξωτερικό Εμπόριο και τη Επιτρόπου Αλίας. Και κάτι άλλο. Το θέμα που πραγματεύεται ο κύριος Καντέκ στην ε, έκθεσή του, το καθεστώς εισαγωγής για τα ελληνικά προϊόντα και τα προϊόντα δετοκαλλιέργειας, θα πρέπει ε, να επικεντρωθεί σε δύο πτυχές. Μία διασταλτική και μία συσταλτική. Σε ό,τι αφορά τη συσταλτική τη συγκεκριμένη, θα πρέπει περιπτωσιολογικά να εξετάζουμε κάθε διαπραγμάτευση, κάθε ξεχωριστή αλληλευτική συμφωνία. Τώρα, ως προς τη διασταλτική πτυχή, την πιο γενική, νομίζω ότι σκόπιμο θα ήταν να υιοθετήσω μια πιο ευρία προοπτική για τα συστήματα εισαγωγής, για το καθεστώς εισαγωγής εν γέννη. Κάτι αντίστοιχο ισχύει στην Επιτροπή Γεωργίας για το κρέας ή άλλα προϊόντα που εισάγουμε. Νομίζω ότι οι αποφάσεις μας για τις συμφωνίες αυτές θα ενισχυθούν αν ενταχθούμε σε μια ευρύτερη πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα εισαγόμενα προϊόντα. Γιατί πολλές από τις πτυχές που επισημάναμε εμεί η χνηλασιμότητα, η πιστοποίηση, ο θεμητό και όχι αθέμητο ανταγωνισμό. η απέτηση να ισχύουν ίδιες συνθήκες παραγωγής στους ντόπιου και στους παραγωγούς τρίτων χωρών. Όλα αυτά τα θέματα ανακύπτουν για όλες τις εισαγωγέ και για τι συμφωνίες που μας ενδιαφέρουν, αλλά και για γεωργικά προϊόντα. Οπότε σκόπιμο θα ήταν να ενταχθούμε σε μια ευρύτερη προοπτική, γιατί έτσι θα ενισχυθεί και η θέση μας ως προς προϊόντα. Αν ενταχθούν αυτά σε μια ευρύτερη κοινή πολιτική που θα καλύπτει όλα τα εισαγόμενα προϊόντα πρώτης ανάγκης που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πατράου. Έχω και εγώ κάποια σύντομα σχόλια. Να συγχαρώ και εγώ τον κύριο Καντέκ για την έκθεσή του και θα ήθελα να επισημάνω δύο-τρία σημεία. Όταν μιλάτε για συγκεκριμένες προτάσεις ε, και λέτε ότι θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται σε θέματα εμπορικών προϊόντων και ο αρμόδιος επίτροπος θα πρέπει να είναι η επίτροπος αλίας. Ε, μου φαίνεται πάρα πολύ καλό, και, αλλά δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουν σε ασχολούνται με το εμπόριο. Εμένα μου φαίνεται εξαιρετικό, διότι πάντα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ε, ενώσεως θέλουμε να ε, αυξήσουμε τα λευτικά προϊόντα. Οι χώρες όπως η Γερμανία ε, εισάγουν τα πάντα για παράδειγμα. Θα πρέπει λοιπόν η ε, δασμοί να είναι και κατάλληλοι για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον κλάδο μας και θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω ε, και αυτό που προσπάθησε να κάνει ο κύριος Λαμή κάθε φορά που έκανε ένα ταξίδι ο κύριος Λαμή ήταν μεγάλη αποτυχία διότι οι δασμοί των ε, ε αλλιευτικών προϊόντων μειωνόντουσαν κατά 50 ή 60% ε, τον τόνο για παράδειγμα. Ε, στην Ταϊλάνδη και στις Φιλιππίνες ε, οι δασμοί για τις ε, κονσέρβες και τα προϊόντα τόνου εν γέννη μειώθηκαν κατά τέτοιο βαθμό που για κάπου αρκετά χρόνια καταστρέφει και ο δικός μας ο κλάδος. Ε, τις ε, τελευταίες ε, εβδομάδες πήγαμε στη χώρα των Βάσκων και διαπιστώσαμε ότι όλη αυτή η πολιτική δεν ήταν καλή για τις περιοχές μας και στην Ταϊλάνδη αυτή τη στιγμή βρίσκονται οι μεγάλες πολυεθνικές οι οποίες εγκαταστάθηκαν μετά από όσα έκανε ο κύριος Λαμή. Και αυτή τη στιγμή όχι μόνο δεν συμμορφούνται και δεν έχουν ε, Ταϊλανδούς υπαλλήλου, αλλά έχουν σκλάβους εντό αγωγικών από την ε, ε, Βυρμανία, τους οποίους ε, πληρώνουν 60 cents την ημέρα και καταλαβαίνετε τι ακριβώς γίνεται εκεί. Αυτά όλα αποτελούν απόδειξη ότι η πολιτική αυτή δεν ήταν καλή. Στην Παππούα Νέα γυναίκα αυτή τη στιγμή πηγαίνουν και κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλες αυτές οι πολιτικές ε, θα πρέπει να είναι στοχευμένες, θα πρέπει να υπάρχουν προτεραιότητες οι οποίες ε, θα πρέπει να βοηθούν την ανάπτυξη μεν, αυτό είναι πάρα πολύ καλό, αλλά δεν θα πρέπει να δημιουργούν προσκόμματα στο δικό μας τον κλάδο και να δημιουργούν και προβλήματα σε τρίτες χώρες όπως αποδεικνύεται. Πολλές φορές ε, γίνονται διαπραγματεύσεις λανθασμένες και αναφέρομαι κυρίως στην εποχή του κυρίου Λαμή. Συμφωνώ λοιπόν απολύτως ότι θα πρέπει ε, οι επίτροποι μας να κάνουν κάτι καλύτερο και να λάβουν υπόψη τα συμφέροντα και των δύο πλευρών. Θα είναι πάρα πολύ εύκολο και για τον κύριο Λαμή και για άλλους επιτρόπους. Δεν θέλω να μιλάσω ε, γιατί δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή και δεν νομίζω θα προσβληθεί για τα όσα λέω. Είναι πολύ εύκολο να έρθουν οι επίτροποι και να λένε κάποια πράγματα χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τις επιπτώσεις που μπορεί να υπάρχουν. Και βλέπετε πόσο αρνητικές ήταν οι επιπτώσεις μετά από τις διαπραγματεύσεις που έκανε ο κύριος Λαμή. Μετά από όλα αυτά λοιπόν να περάσω σε ένα άλλο θέμα, το θέμα του ΠΟΕ. Συμφωνώ απολύτως ότι το θέμα των επιδοτήσεων το οποίο συζητάτε, η επιδοτήση της, επιδότηση επιδοτήσεις κοινωτικής πολιτικής ε, στον αλληλευτικό τομέα, ε, είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί και θα πρέπει να μειωθούν οι επιδοτήσεις. Εγώ είμαι από τους πρώτους, παρόλο που κάποιοι θεωρούν ότι εγώ δεν προασπίζομαι αυτά τα θέματα που τα προασπίζομαι. Υπάρχει όμως και το αντίβαρο εδώ. Και δεν θα πρέπει να επιμείνουμε σε κάποιες πολύ συγκεκριμένε ε, πτυχές. Θα πρέπει να τονίσουμε, για παράδειγμα, το θέμα της απελευθέρωσης των επιδοτήσεων. Διότι εδώ όλοι θέλουν να μειωθούν οι επιδοτήσεις, αλλά εγώ θα πρέπει, πιστεύω ότι θα πρέπει να απελευθερωθούν οι επενδύσεις, όπως κάναμε γενικότερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά την οικολογική σύμβαση, εγώ συμφωνώ, ήμουνα και εισηγήτρια στο θέμα της οικολογικής σήμανσης και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τηρεί τις υποχρεώσεις που ανέλαβε. Και θα ήθελα εδώ να τραβήξουμε ταυτή μόνο, όχι μόνο όσους ασχολούνται με το εμπόριο, αλλά και όσους ασχολούνται με την αλία. Δεν συμφωνώ 100% με τα όσα γράφεται για τις ε, ε σημάνσεις. Ε, δεν είναι όλοι άγιοι και δεν είναι όλοι άμυροι ευθυνών υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι ε, εμπορεύονται προϊόντα τα οποία είναι πάρα πολύ ακριβά και ε, δεν είναι τόσο ε, δεν έχουν τόσους εκβιασμούς, αλλά και πάλι ε, αυξάνουν πάρα πολύ τις τιμές. Θα πρέπει να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι στόχοι οι οποίοι θα είναι αντικειμενικοί και θα, που θα χρησιμεύσουν πραγματικά σε οικολογική σήμανση. Θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάποια θέματα κοινωνικού ντάμπινγκ κλπ. Αλλά επειδή μας πιέζει ο χρόνος να δώσω απευθεία το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, τον κύριο Σωμόζη, ελπίζω να μην ε, σας επηρεάζουν εσά οι επικρίσεις που έκανα, αλλά θα ήθελα η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου να προασπίσει τον εαυτό της και όχι μόνο ο κ. Λαμή που δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή, αλλά θα ήθελα να προασπίσετε τον εαυτό σας για τις θέσεις που ακούσαμε ε, βάσει της έκθεσης του κ. Καντέκ. Παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου εκπρόσωπος της Επιτροπής. Ε,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 Τώρα έχω το μικρόφωνο και ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για το που μου δώσετε το λόγο και ευχαριστώ και τον κύριο Καντέκ για το πολύ ενδιαφέρον έγγραφο εργασίας. Είχαμε μία σύντομη συζήτηση πριν από τη συνάντηση αυτή και στην αρχή ο κύριος Καντέκ είπε ότι είναι απλώς ένα έγγραφο εργασίας για να μας ε, οθήσει να σκεφτούμε και να σημειώσουμε ορισμένες αντιδράσεις ε, των Ευρωβουλευτών ή των ε, ενδιαφερομένων του κλάδου. Ε, πρέπει να συζητηθεί πολύ σοβαρά στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι μιλώ εν ονόματι της Γενικής Διευθύνσεως Εμπορίου. Υποθέτω ότι υπάρχουν συνάδελφοι από την Γενική Διεύθυνση Θαλάσσης, την DG Mare, που ίσως έχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά θα ήθελα να τονίσω επίσης ότι ακόμη ε, προσπαθούμε να χωνέψουμε το έγγραφο αυτό, ιδίως όσον αφορά τις, ε, τα σχόλια για τις εσωτερικές ε, ευθύνε που πρέπει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναλύουμε και τις ανησυχίες σας σχετικά με το κεφάλαιο σχετικά με τις ε, ε, εμπορικές διαπραγματεύσεις. Ε, κυρία Πρόεδρε, έχω μία γραπτή δήλωση η οποία ε, έχει το πράσινο φως της Γενικής Διεύθυνσής μου και θα ήθελα να την διαβάσω. Θα διατηρήσει 5-6 λεπτά σχετικά με την πολιτική μας στα πλαίσια αυτού του εγγράφου. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Έχετε πέντε λεπτά να τη διαβάσετε, αλλά πραγματικά με ξενίζει το γεγονό ότι δεν έχετε την ειλικρίνεια να απαντήσετε σε συγκεκριμένε ερωτήσει που διατυπώθησαν για θέματα που αφορούν τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Μπορείτε βέβαια να διαβάσετε ένα κείμενο αν θέλετε, είστε ελεύθερο να κάνετε ό,τι θέλετε. Εμένα δεν μου φαίνεται σωστό από πλευρά Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Καταλαβαίνω ότι η επίκριση δεν είναι προ εσά που είστε ένα υπάλληλο απλώ. Σα δίνω λοιπόν τα πέντε λεπτά να διαβάσετε αυτό που θέλετε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Βέβαια, η έκθεση αυτή θα αναφέρεται στα περισσότερα ερωτήματα και σχόλια τα οποία έχουν θυγεί από τον εισηγητή και ε, από τα σχόλια από τα μέλη της Επιτροπής. Αναφερόμαστε στην έκθεση κατά πρωτοβουλία διότι κατά τη συζήτηση σχετικά με το ρόλο της, ε, του τομέα της αλληλείας πρέπει να ε, τονίσουμε ότι τα ε, θέματα επηρεάζονται από την ε, αναθεώρηση της κοινή πολιτικής αλληλείας ε, και θέματα ανάπτυξης. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι βασικό να λάβουμε υπόψη μερικά βασικά στοιχεία σχετικά με την με την με τον τομέα αυτό. Και ε, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ευθύνεται για την ε, αρμονική εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου και την μείωση των δασμών και άλλων εμποδίων που προβλέπονται από τις συνθήκες Λισαβόνα Λισαβόνας και τις προηγούμενες. Όπως αναφέρεται στις συνθήκες, η κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της γενικής εξωτερικής πολιτικής της Ενώσεως και γι' αυτό εκτός από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 προάσπιση των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως υπάρχουν και άλλα θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως παραδείγματος χάρη οι ευθύνε έναντι των υποανάπτυξη χωρών διότι προβλέπεται ότι στις περιοχές ελευθέρου εμπορίου τα, οι δασμοί και άλλα εμπόδια θα εξαλειφθούν και ε, θα μπορέσει να υπάρξει μια, ένας ενιαίος χώρος Σύμφωνα όμως με τις προτιμησιακές μας συμφωνίες προσπαθούμε να επιτύχουμε μία ισοσκελισμένη και εναρμονισμένη μείωση των δασμών χωρίς να σημαίνει ότι θα εξαλειφθούν όλοι οι δασμοί. Ε, η εξάλληψη των προστατευτικών δασμών δεν θα είναι άμεση ούτε θα είναι ο τελικός στόχος της κοινή εμπορικής πολιτικής. Ε, σαν γενική διεύθυνση για την εμπορική πολιτική εξετάζουμε όλους τους τομείς. Πράγμα το οποίο σημαίνει ε, ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεκτική αντιμετώπιση ε, όλων των πολυμερών και διμερών συμφωνιών στην προετοιμασία των θέσεών μας ε, και ε, μία ε, αντίφαση μεταξύ διαφόρων γενικών διευθύνσεων θα ήταν αρνητική. Δεν σημαίνει αυτό ότι κινούμεθα μόνοι μας, προσπαθούμε να ευθυγραμμιστούμε εις την εξωτερική πολιτική, αλλά συνεργαζόμαστε και στην εσωτερική πολιτική που καλύπτουν τους διάφορους εμπορικούς τομές, μάρε, περιβάλλον, επιχειρήσεις και με τους ενδιαφερόμενους και τα κράση μέλη ούτως ή άλλως δίδουν τις κατευθυντήριες γραμμές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προβεί ε, σε διαπραγματεύσεις και κατά τη διαδικασία αυτή η Επιτροπή ενημερώνει και το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προσπαθούμε λοιπόν να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υπάρχει κι άλλο ένα θέμα το οποίο έχει σχέση με τη μορφή των ε, εμπλεκομένων προϊόντων διότι υπάρχουν ε, αντικρώμενα συμφέροντα μεταξύ των αλληλευτικών προϊόντων της γεωργίας και των εμπορικών μεθόδων κατόπιν ε, του γύρου της Ουρουγουάης προηγουμένως όλα τα γεωργικά προϊόντα δεν μπορούσαν να υποστούν μειώσεις ενώ υπήρξαν έκτοτε στρεβλώσεις στην παγκόσμιο αγορά ε, των γεωργικών προϊόντων και θα πρέπει αυτά τα προϊόντα να εξετάζονται ε, χωριστά και να υπάρξει μία νέα συμφωνία. Η ίδια αντιμετώπιση βασίστηκε εις τις διαπραγματεύσεις ε, για πολλά θέματα, για ε, ευαίσθητους τομείς, ε, για τα χημικά, τις χημικές ουσίες, για τα κλωστοεφαντουργικά και το καθεξής. Γι' αυτό και συνεργάζονται οι διάφορες γενικές διευθύνσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής και όσον αφορά την κοινή πολιτική γεωργίας Αλίας ε, μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, ξεκινήσει διαπραγματεύσεις σχετικά με τις δασμολογικές αλλαγές κατά τρόπον ώστε να ε, μπορέσει η Ευρώπη να παραμείνει ανταγωνιστική χωρίς να βασίζεται μόνο εις τους δασμούς που θα πρέπει ούτως ή άλλως στο μέλλον να μειωθούν. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να σεβαστεί τι τις ε, πληροφορίες ε, του εισηγητή όσον αφορά την κατάρτιση της εκθέσεώς του και έτσι ελπίζουμε ότι ε, θα βελτιώνονται και στο μέλλον οι σχέσεις μας με την, την αντιπροσωπεία σας. Ο, ο κύριος Ραμπό από τη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας καθησυχάζω ότι εγώ δεν πρόκειται να διαβάσω καμία δήλωση. Θα προσπαθήσω να είμαι σχετικά λακωνικός. Εκπροσωπώ τη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσης και κυρίως ε, την Γενική Διεύθυνση Αλίας και Θάλασσης εκπροσωπώ και ίσως υπάρξει μια διαφοροποίηση σχέση με αυτά που ακούσαμε προηγουμένως. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν το έγγραφο αυτό είναι πλήρες και διεξοδικό σε ό,τι αφορά τα διάφορα, τις διάφορες πλευρές ε, του εμπορίου για, την, για τα ελευτικά προϊόντα και την υδατοκαλλιέργεια. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της έκθεσης αυτής που επιδοκιμάζουμε ιδιαίτερα είναι ότι προβαίνει στην υποβολή κάποιων λύσεων και προτάσεων σε ό,τι αφορά τις πρακτικές των τελευταίων ετών για τα λευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας. Τώρα, υπό το πρίσμα της κοινή ελευθερίκης πολιτικής, αυτή η έκθεση είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη και πολύ επίκαιρη, γιατί υποβάλλεται τη στιγμή που έχουμε ξεκινήσει μια μεταρρύθμιση της κοινή ελευθερίκης πολιτικής και του σκέλους της κοινή οργάνωσης αγορών. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε τέσσερα βασικά στοιχεία της έκθεσης που αναφέρθηκαν το πρωί και αφορούν καταρχήν τα εμπορικά εργαλεία, τους εμπορικούς μηχανισμούς. Αυτά τα εργαλεία, αυτοί οι μηχανισμοί θα ρυθμίσουν τις ροές κυρίως από τις τρίτες χώρες, τις εισαγωγές από τις τρίτες χώρες. Στο μέτρο που έχουμε μια δασμολογική πολιτική με συγκεκριμένους κανόνες. Όταν θα καταργηθούν ε, τα τέλη και οι δασμοί, δεν θα χρειαζόμαστε καν τέτοιους ε, μηχανισμούς ρύθμισης όπως είναι η αναστολή για παράδειγμα, όπως αναφέρει η έκθεση Καντέκ. Αναφέρονται και άλλα εργαλεία όπως είναι η υγειονομική έλεγχη. Το έχουμε ξανασυζητήσει και εδώ, αλλά αναφέρεται και σε άλλες περιπτώσεις ε, και είναι χιλιοσυζητημένο το θέμα των υγειονομικών ελέγχων. Έχουμε ένα σύστημα προστασίας της υγείας του καταναλωτή που είναι το καλύτερο στον κόσμο. Οπότε δεν θα πρέπει να υπονομεύσουμε ή να διακυβεύσουμε αυτό το σύστημα. Ίσως, αν χρειαστεί, αν παραστεί ανάγκη, καλό θα ήταν να επιτείνουμε τους ελέγχους στα εισαγόμενα προϊόντα. Πάντως, το ίδιο το σύστημα επουδενή δεν πρέπει να αφισβητηθεί. Ένα άλλο σύστημα ελέγχου για τα εισαγόμενα προϊόντα ε, προκύπτει από το νέο κανονισμό για την πάταξη της παράνομης αλίας και νομίζω ότι είναι Πολύ χρήσιμο αυτό το σύστημα πιστοποίηση που εγγυάται ότι τα αλληλευτικά προϊόντα, όχι τα προϊόντα του καλλιέργεια, αλλά τα αλληλευτικά προϊόντα που εισάγονται στην Ένωση θα πρέπει να έχουν προηγουμένω στηρίσει όλου του ε, κανόνες, ε, τους συντήρηση. κανόνες συντήρησης. Τρίτο στοιχείο που αναφέρθηκε πολλάκι είναι η ιχνηλασιμότητα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αν θέλουμε να ενημερώσουμε τον ε, καταναλωτή πλήρως για να έχει εμπιστοσύνη στο προϊόν που καταναλώνει, που αγοράζει. Ο περσινός νέος κανονισμός ελέγχου θέσπισε ένα τέτοιο νέο σύστημα και προσπαθούμε να εφαρμόσουμε κάποια εκτελεστικά μέτρα για τον κανονισμό αυτό. Πάντως αυτό το σύστημα, αυτός ο κανονισμός θα προβλέψει τα απαραίτητα εχέγγυα και για τα εισαγόμενα προϊόντα, για σωστή και διεξοδική ενημέρωση του καταναλωτή. Κύριε Πρόεδρε, εσείς έχετε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό και το επισημάνατε, είναι πολύ σημαντικό. Είναι το θέμα της σήμανσης ή της οικολογικής σήμανσης ή ετικετοθεσίας. Νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία τη μεταρρύθμισης τη κοινή αλληλευτικής πολιτική. το θέμα των πληροφοριών που χορηγούνται στον καταναλωτή για τα αλληλευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας. Αυτή τη στιγμή ισχύουν κάποιοι κανόνε που θεσπίζουν υποχρεώσει σήμανση για τα αλληλευτικά προϊόντα. Είναι απλούστατοι οι κανόνε αυτοί και από ό,τι φαίνεται ανεπαρκείς, γιατί δεν ενημερώνουν σωστά τον καταναλωτή. Αλλά και οι υπόλοιποι φορεί του κλάδου δεν είναι πολύ ικανοποιημένοι. Οπότε θα πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση αυτής της ενημέρωσης. Καλό θα ήταν οι οικειοθελείς πληροφορίες που μπορούν να συνοδεύουν ένα λευτικό προϊόν και ε, προϊόν υδατοκαλλιέργειες να πλαισιωθούν. Για παράδειγμα, κάποιοι ισχυρισμοί που αφορούν το περιβάλλον ή το γεγονό ότι εφαρμόστηκαν μέθοδοι αηφόρου αλεία για την αλεία του συγκεκριμένου προϊόντο. Πάντω, στη μεταρρύθμιση αυτή θέλουμε ένα ευρύ πεδίο ένα ευρύ φάσμα, ώστε στο μέλλον να καλύψουμε οποιοδήποτε ισχυρισμό, οποιοδήποτε μνήα που μπορεί να συνοδεύει ένα λευτικό προϊόν, προκειμένου ο καταναλωτής να ενημερώνεται σοβαρά και διεξοδικά για να προβεί σε μια, σε μια ε, υπεύθυνη αγορά και κατανάλωση. Αυτά κύριε Πρόεδρε και είμαστε στη διάθεσή σας. Και μία άλλη πληροφορία, γιατί ρωτήθηκε το κατά πόσο εισαγωγέ καλύπτουν την παραγωγή κοινοτικών σκαφών στα πλαίσια των αλληλευτικών συμφωνιών. Η απάντηση είναι αρνητική γιατί τα προϊόντα αυτά θεωρούνται κοινοτικά προϊόντα. Και αν θυμάμαι καλά, η παραγωγή των κοινοτικών σκαφών στα πλαίσια των αλληλευτικών συμφωνιών καλύπτουν ένα 10% όχι του συνολικού ανεφοδιασμού, αλλά 10% του κοινοτικού ανεφοδιασμού. Ευχαριστώ. Ε, ε, Ευχαριστώ. Ο κύριος Καντέκ για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι διότι συμμετείχατε τόσο ευραίως σε αυτή την πρώτη ανταλλαγή σχετικά με το έγγραφο εργασίας, πράγμα που δείχνει πόσο σας ενδιαφέρει. Πιστεύω λοιπόν ότι χάρη στην συνδρομή σας θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μία πιο συγκεκριμένη έκθεση που να αντιπροσωπεύει αυτό το οποίο εσείς σκέφτεστε. Δεν θα απαντήσω μεμονωμένα στον καθένα από εσά, αλλά σύντομα ε, ορισμένες παρατηρήσεις. Ε, σχετικά με τις συμφωνίες ε, εισαγωγής σας απάντησε η Γενική Διεύθυνση Θαλάσσης. Όσον αφορά την ρήτρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βεβαίως πρέπει να τις σεβαστούμε. Στρούαν αναφέρθηκε ιδίω στην υδατοκαλλιέργεια. Νομίζω ότι είναι ένα τομέα στον οποίο επεξεργάζεται ο συνάδελφος Μιλάνα, ο οποίος θα επανέλθει στο θέμα αυτό και για το παγκάσιο και για τα προϊόντα που προέρχονται από την Νορβηγία. Αλλά όπως όλοι εδώ ε, πρέπει να υπάρξει ε, μια υγειονομική δικαιοσύνη μεταξύ όλων των προϊόντων ευρωπαϊκών μη εισαγωμένων δηλαδή. Ε, θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα κοινοτικό προϊόν το οποίο σημαίνει ότι έχει αλλιευθεί εντός ε, εντός των υδάτων της ενώσεως από πλοίο ε, κοινοτικό ή εκτός των ε, υδάτων της ενώσεως από πλοίο με κοινοτική σημαία για να είμαστε συνεννοημένοι. Νομίζω ότι αυτά, σε αυτό συμφωνούν όλοι. Υπάρχει και το, η ευρωπαϊκή σήμανση. Θα πρέπει να προσέξουμε τα, τις ιδιωτικές σημάνσεις οι οποίες ακολουθούν ατάκτους ε, ε, ε, οδούς. Θα ήθελα λοιπόν όσον αφορά τις τεχνικές ερωτήσεις σου να σου απαντήσω λίγο πιο συγκεκριμένα διότι αναφέρονται σε πολλά σημεία μιλώ προς την κυρία Λέβιν Μιλήσαμε και για τα θέματα των καυσίμων, αλλά αυτό ε, στα περιθώρια της σημερινή μας συζητήσεως. Γενικώ όμως νομίζω ότι και τα δικά σας σχόλια ήταν πολύ σημαντικά. Ο κύριος Φερέρα μας ξαναείπε και δεν μας κατέπληξε την αντίθεσή του σε κάθε απελευθέρωση, το αντιλαμβανόμαστε, δεν περιμέναμε το αντίθετο, αλλά πρόκειται για σχόλια ε, ε, καταληκτικά και στην αρχή προσπάθησα να είμαι πολύ πιο προκλητικός διότι υπάρχουν συγκρόμενα συμφέροντα όπως το είπατε και πρέπει να το τονίσουμε, πρέπει να το προσέξουμε διότι επηρεάζει όλες τις προτάσεις τις οποίες μπορεί να διατυπώσουμε. Κύριε Μιλάνα. Εσείς μου μιλήσατε για τα κοινοτικά προϊόντα, όπως είπαμε, και επίσης αναφέρθηκε στον εντοπισμό της ευρωπαϊκής παραγωγής. Ε, ε, θα μου γράψεις κάτι, θα το περιμένω βεβαίως ε, και μη διστάσει και όποιος άλλος θέλει να μου στείλει σημειώσεις όταν είπαμε πώς θα ενταχθεί η σκέψη αυτή στην πράσινη βίβλο είναι βέβαια δύσκολο διότι είναι τεράστια η πράσινη βίβλος αλλά θα προσπαθούσαμε να το ενσωματώσουμε. Ο κύριος Βάρια μας είπε ότι το θύμα είναι πολύ περίπλοκο και γι' αυτό μας απασχολεί και είναι θέμα αγοράς. Η αγορά είναι μια ενιαία αγορά και ε, η επίπτωση κάθε εισαγωγικής συμφωνία στην αλληλεία είναι κάτι το οποίο επίσης θα τροφοδοτεί στην έκθεση αυτή. Με μεγάλη χαρά άκουσα ότι ο συνάδελφος από τη Φιλανδία ε, ε, ψάρευε το Σαββατοκύριακο στο Πάγο, μάλλον κάτω από τον Πάγο και θα ήθελα μια φορά να πάμε στη Φιλανδία να μας το δείξει αυτό, διότι πιστεύω ότι το καλύτερο ψάρι είναι το φρέσκο ψάρι, το νοπό ψάρι. Ε, και αυτό είναι πολύ φρέσκο με όλη τη σημασία της λέξης εφόσον είναι κάτω από τον πάγο. Ε, αυτό μας οδηγεί στη σήμανση και νομίζω ότι όλοι το επανέλαβαν ότι το θέμα αυτό βρίσκει σύμφωνη όλη την Επιτροπή. Η Μαρία Πατράης μας είπε ότι δεν επαρκούν οι καλές προθέσεις, θα πρέπει να καταλήγουν σε συγκεκριμένα μέτρα και πιστεύω ότι όλοι το αντελήφθησαν. Βέβαια δεν συμφωνούμε όλοι πλήρως σχετικά με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ή της Επιτροπής Αλληλείας σχετικά με τα αλληλευτικά προϊόντα. Έχω μία άποψη την οποία συμμερίζεται η Κάρμεν αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν κι άλλες μπορούμε να το συζητήσουμε. Και ε, γι' αυτό τόνισα και αυτό το θέμα. Επίσης ε, όσον αφορά την ε, χειμερινή αντιμετώπιση, ο, ο Πασκάλ Λαμή είναι έτοιμος για τα δύσκολα, με χειμερινή ένδυση δηλαδή, ε, ενδυμασία και ε, η Κάρμεν ε, θύμισε ε, ε, τη σημασία της οικολογικής σήμανσης τονίζοντας ορισμένες πιστοποιήσεις που ήδη υπάρχουν και εγώ συμφωνώ για την απελευθέρωση των επενδύσεων που μας απασχόλησε επίσης. Θέλω όμως να ευχαριστήσω τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και για τις ανταλλαγές τις οποίες είχαμε πριν από την κατάρτιση του εγγράφου αυτού, διότι κατόπιν ανταλλαγών με τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου καταλήξαμε στο κείμενο αυτό και τους ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μας έδωσαν, αλλά εκπλήσωμε όπως και η πρόεδρος η Κάρμεν να χρειαστεί ένα γραπτό κείμενο αντί για απάντηση σε ορισμένες ερωτήσεις. Θα σας υπενθυμίσω όπως είπατε και εσείς ότι η συνθήκη της Λισαβόνας δεν είναι μόνο η ανάγνωση όλων των άρθρων της συνθήκης αλλά ιδίω κατά τη γνώμη μου μια νέα ισορροπία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καλύτερα λοιπόν να επαναλαμβάνουμε για να μην διαφωνούμε όπως έλεγαν οι Έλληνες ε, θα επαναλάβουμε και λέμε ότι η συνθήκη τη Λισαβόνας υπάρχει σήμερα και αυξάνονται οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε επίσης λόγο για την μελλοντική ανάπτυξη της αλληλείας. Ευχαριστώ τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ για τη συνδρομή της αυτό το έγγραφο εργασίας και για τη στήριξή της, την ουσιαστική στήριξή της στο έγγραφο αυτό με ορισμένες παρατηρήσεις τις οποίες θα περιλάβω όσον αφορά τα εμπορικά εργαλεία. Όπως παραδείγματο χάνει, όπως ανέφερα, τους ελέγχους για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας από την Άπο αλλά θα χρειαστεί να πολλαπλασιαστούν οι έλεγχοι αυτοί αν έχουμε τις δυνατότητες, διότι οι εστιασμένες επεμβάσεις πολλές φορές δεν επαρκούν και επίση τον έλεγχο τη παράνομη αλληλεία και την εχνηλασιμότητα που αποτελεί ένα βασικό στοιχείο όπως και η σήμανση. Ευχαριστώ ε, όλους για αυτέ τι ανταλλαγέ, για αυτή την ανταλλαγή η οποία ήταν πολύ πλούσια. Περιμένω τα γραπτά σας σχόλια για να μπορέσω να τροφοδοτήσω περαιτέρω την έκθεση αυτή και ευχαριστώ την Πρόεδρο που μου έδωσε τη δυνατότητα να παρουσιάσω σήμερα αυτή την έκθεση και όλους τους συναδέλφους από όλες τις ομάδες. Εγώ ευχαριστώ κύριε Καντέκ. Ήσασταν και τυχερόν για... τυχερός γιατί ήταν ε, σχετικά άδικο το πρωινό, επομένως μπορέσαμε να έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Σομιγή από τη Γενική Διεύθυνση Trade και τον κύριο Ραμπό. Επιμένω να μην πάρετε προσωπικά τα σχόλια ε, που ακούσαμε κάποιες επικρίσεις ε, από πλευράς Γενικής Διεύθυνσης Trade δεν ε, θέλουμε να επιτεθούμε στους υπαλλήλους αλλά σε, στους ηθήνοντες της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής που δεν σκέφτονται αυτό που θα έπρεπε να σκέφτονται και στέλνουν τους υπαλλήλους εδώ να δεχθούν τα πειρά. Να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης και επειδή θα γίνει και κλεισμένο των σειρών θα ήθελα να ζητήσω εκτός από τους Ευρωβουλευτές και τη Γραμματεία της Επιτροπής Ελίας και τη Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι υπόλοιποι παρακαλώ να αποχωρήσουν για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ.